επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Ε, είναι καλό πάντοτε τους πόρους μας που είναι τόσο λιγοστοί και πολύτιμοι να τους χρησιμοποιούμε με τον πιο φιδωλό τρόπο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κάλανα. Να έχει κλείσει και αγαπητοί συνάδελφοι η συζήτηση. Ψηφοφορία αύριο στι 12. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι αυτό του κυρίου Κάντσαν για το δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Καλώς ήρθατε. Κύριε Γκόρν, κύριε Επίτροπε Κάλλας, κύριε Καντσάν, τέσσερα λεπτά. Οι διαπραγματεύσεις που ανέλαβα κατά το πρώτο έτος μόνος μου και στη φάση συνδιαλλαγής, για την πρώτη συνδιαλλαγή μετά την συνθήκη της Λισαβόνας, με την βοήθεια της κυρίας Κράτσα Τσανκαροπούλου και την υποστήριξη του Προέδρου της Επιτροπής ε, Τουρισμού, του κυρίου Σίμψον, ε, οδήγησε σε αποδεκτά αποτελέσματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα 70 εκατομμύρια επιβατών θα έχουν ε, μια σειρά δικαιωμάτων που σήμερα ήταν ανύπαρκτα εάν τα συγκρίνουμε με άλλους τρόπους μεταφοράς. Οι στόχοι που θέσαμε με βάση τις τρεις προεδρίες ήταν ε, οι εξής. Ένας κανονισμός ο οποίος να εποπτεύει τις μη διακρίσεις κατά την μεταφορά με πούλμαν ή λεωφορεία, να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα όπου απασχολούνται ΜΜΕ που δεν μπορούν να έχουν περαιτέρω επιβαρυνσεις. Επίσης να καλύψουμε ένα ρυθμιστικό κενό που υπήρχε στον τομέα των λεωφορείων και των πούλμαν σε σχέση με άλλους τρόπους μεταφοράς για να υπάρχουν ελάχιστες εγγυήσεις για όλους τους επιβάτες. Επίσης ένα κανονισμό ο οποίος να ε, βοηθήσει τα τα δικαιώματα των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στα πλαίσια της γύρανσης του πληθυσμού αυτά τα μέσα θα χρησιμοποιούνται όλα ένα και περισσότερο, γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε και τα δικαιώματα αυτής της κατηγορίας. Τα βασικά προβλήματα ανέκυψαν στον ορισμό του πεδίου εφαρμογής. Κύριε Καντσάν μπορείτε να μειώσετε την ταχύτητά σας, διότι δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε αφορούν τον ορισμό του πεδίου εφαρμογή, διότι ο κανονισμός ισχύει σε ε, ε, εθνικό διασυνοριακό επίπεδο, περιφερειακό και τοπικό για μια απόσταση που υπερβαίνει τα 250 χιλιόμετρα. Μιλάμε για βασικά δικαιώματα τα, για τα οποία ισχύει αυτό το όριο. Μιλάμε για το δικαίωμα μεταφοράς, την ε, κατάσταση, την, κατάρτιση, την πληροφόρηση και την ευθύνη που φέρει ο, ο δικός φορέας. Ε, πάνω από τα 250 χιλιόμετρα λοιπόν που διανύονται θα πρέπει να υπάρχει αποζημίωση καθώς και ε, αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος και αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης. Επίσης, αποζημίωση για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα αυτές τις υποχρεώσεις του φορέα και θα πρέπει να καταβληθούν μέσα σε τρεις μήνες μετά από την προσφυγή. Επίσης, θα πρέπει να οριστεί ένας νέος φορέας, ο οποίος να είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να παρεκκλίνουν για μία περίοδο τεσσάρων ετών που θα μπορέσει να επαναληφθεί μία μόνο φορά μετά από από κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλούνται τα κράτη-μέλη να ορίσουν ένα ενιαίο εισιτήριο για κάθε φορέα μεταφοράς και για κάθε μέσο μεταφοράς. Το τελικό κείμενο θα είναι ένα κείμενο συμβιβασμού το οποίο είναι ικανοποιητικό. Πιστεύω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία αυτή η διαδικασία συνδιαλλαγής για το Κοινοβούλιο. Τώρα δίνω το λόγο στην ε, κυρία Γιουερή, η οποία θα μιλήσει εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, μεγάλη χαρά συμμετέχω σε αυτή την συζήτηση σε μια πρόταση για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των επιβατών δηληφοριών και πούλμαν για την τροποποίηση του σχετικού κανονισμού. Είναι κατάλληλη στιγμή για την οποία έρχεται η συζήτηση αυτή, ύστερα από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων. Εκ μέρου του Συμβουλίου, καταρχά, θέλω να εκφράσω τι ευχαριστίε μου και την εκτίμηση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία, το πνεύμα συμβασμού που επέδειξε και που μα επέτρεψε να καταλήξουμε συμφωνία στην ε, Επιτροπή τη Συνδιαλλαγή προ ε, το συμφέρον των επιβατών, λεωφορείων και πούλμαν και ιδιαίτερω των ατόμων με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα. Οι συζητήσει μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων δεν ήταν πάντοτε πρόσκοπτε, όμω ήταν πάντοτε επικοδομητικέ και τι καθοδηγούσε συμβαστικό πνεύμα. Το κοινό κείμενο στο οποίο καταλήξαμε με το οποίο καταλήξαμε συμφωνία στην Επιτροπή Συνδιαλλαγή και το οποίο ελπίζουμε θα εγκριθεί σήμερα αποτελεί συμβιβασμό που ικανοποιεί όλε τι πολιτικέ ομάδες. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω τη σοφόρο σε όλους όσοι συνέβαλαν στο σημαντικό αυτό έργο και την ομοθετική πρόταση, ιδιαίτερα στον αντιπρόεδρο, την αντιπρόεδρο κυρία ε, Κράτσα Τζεγκαροπούλου, τον ε, πρόεδρο κύριο Μπράιαν Σίμψον τη Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, τον εισηγητή κύριο Καντσάν και του κοιόδη εισηγητά για τη δουλειά του γιατί όλοι μαζί συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτής της νομοθετικής διαδικασίας και την προαγωγή της σε οικοδομητικό αποτέλεσμα. Τον κύριο Κάλλας επίσης και το επιτελείο του θα ευχαριστήσω καθώς ε, και το προσωπικό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ε, ακαταπώνητοι βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Εν τέλει θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαρισίες μου στη Βελγική Προεδρία για την εξαίρετη δουλειά τη που μα προσέφερε την απαραίτητη στήριξη και μέσα στο Συμβούλιο στις διαδικασίες τη συνδιαλλαγή. Το κοινό αυτό κείμενο που αποτελεί αποτέλεσμα καρπό των εργασιών της συνδιαλλαγής πιστεύω ικανοποιεί πλήρω τα μελήματα για την προστασία των συμφερόντων των επιβατών, πούλμαν και λεωφορείων, ταυτόχρονα διαφυλάσσοντα και τα συμφέροντα των μεταφορικών επιχειρήσεων που είναι επιτοπλίστων μικρομεσαίε. Θέλουμε δηλαδή και σεβασμό των δικαιωμάτων των επιβατών όσον αφορά αποστάσεις έως 250 χιλιόμετρων και εγγυήσεις ε, για τους επιβάτες, για τα δικαιώματα των επιβατών ανάλογα με την απόσταση που διανέουν. Επίσης, ε, άτομα με αναπηρία ή επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα έχουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εξασφαλίσαμε αμοιβαία αποδεκτέ λύσεις για αρκετά δύσκολα ζητήματα. Καταρχάς, το πεδίο εφαρμογή, κατά δεύτερον, τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση καθυστερήσεω ή ματαιώσεω ταξιδιού, ε, στήριξη και βοήθεια, πρώτε βοήθειε σε περίπτωση ατυχήματο, μετάβαση στου νέου κανόνε και εν τέλει τα δικαιώματα των ε, επιβατών με αναπηρία ή με περιορισμένη κινητικότητα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, όπω γνωρίζετε, το Συμβούλιο υιοθέτησε το κοινό κείμενο στι 31 Ιανουαρίου στη συνεδρίασή του. Πρόκειται για ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο μπορεί να υπογραφεί αύριο. Η δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται για τον Μάρτιο. Και ως τελευταία λόγια, συγχαρητήρια στον ε, κύριο Κατσάρ για την εξαιρετική δουλειά του και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ όλους για την ε, πολύ καλή αυτή δουλειά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Αγγιαρή. Ο Επίτροπος ε, Κάλλας τώρα, πρόεδρε. Αξιότιμη συγητά, κύριε Γκέτσεν, κυρία Γκέρι, Πρόσωπε του Συμβουλίου, αξιότιμοι βουλευτές, Η πρόταση για τα δικαιώματα των επιβατών ε, Πούλμαν και λεωφορείων, το θέμα που συζητούμε σήμερα δηλαδή, είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης ε, διαδικασίας ε, και συνδιαλλαγής μακρές διαπραγματεύσεις μέχρι αργά τη νύχτα, θυμηθείτε τον Νοέμβριο την Επιτροπή συνδιαλλαγή και τελικά μετά από πάνω από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων καταλήξαμε σε συμβαστική λύση επιτέλους. Σας ευχαριστώ θερμά για τις προσπάθειές σας ε, κυρία Κράτσα πρώτα απ' όλα για, την για τον ηγετικό σας ρόλο και προς τον κύριο Σίμψον, προς τον κύριο Κάντσαν, τον εισηγητή και προφανώ να ευχαριστήσουμε και την ε, Βελγική Προεδρία. Είμαι ευγνώμων προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι ανέκαθεν επιζητούσε μια ισχυρή ε, μεγάλη προστασία των επιβατών. Στη, την 31η Ιανουαρίου κατέληξε σε εκνηθέ στο Συμβούλιο και σα καλώ να εγκρίνετε κι εσεί ε, την πρόταση και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οι επιβάτε των Πούλμαν και Λεωφορείων ε, ε, έχουν τώρα μία πλήρη προστασία και τα μέτρα είναι ποφελή για τους καταναλωτές και κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών όπου και αν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συμβαστικό κείμενο ε, περιέχει σημαντικά επιτεύγματα, μία σειρά βασικών ε, οικουμενικών δικαιωμάτων για όλους όσους μετακινούνται με πούλμαν και λεωφορείο. Φυσικά, όπως είπε ήδη ο κύριος Κάντσον, υπάρχουν και κάποια επίμαχα αμφιλεγόμενα ζητήματα που ε, γύραμε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων σχετικά σχετικά με το πλαίσιο του κανονισμού. Συγκεκριμένα η απόσταση από 250 χιλιόμετρα και πάνω ε, θεωρείται ότι είναι υπερβολικά μεγάλη απόσταση και θέλετε να προστατευτούν και οι τοπικές μετακινήσεις. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι η εφαρμογή των διατάξεων επιφέρει μεγάλο κόστος κυρίως για τους μικρούς μεταφορείς. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ίσως κελισμένη, μια ισόρροπη πρόταση. Μην ξεχνούμε ότι τα βασικά δικαιώματα προβλέπονται για διάφορα είδη υπηρεσιών και παρέχουν ιδιαίτερη προστασία για τους ευάλωτους ευπαθείς επιβάτες. Επίσης, ε, το κόστος ε, για την βιομηχανία προσπαθούμε να το διατηρήσουμε σε ελάχιστα επίπεδα συνολικά. Το συμβαστικό κείμενο συνιστά ένα άλμα, μια πραγματική πρόοδο και για τους επιβάτες και για την εικόνα της ε, βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Θα ακούσουμε τώρα τους ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Γκρός, εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αγαπητοί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα στον κύριο Καντσάν, τον συνάδελφο, για τη συνεργασία. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το θέμα που είχαμε να συζητήσουμε και που φέραμε σε αίσιον πέρα, πιστεύω. Βεβαίω, οι συμβασμοί πάντοτε έχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Για άλλου είναι υπερβολικοί, για άλλου είναι μινιμαλιστικοί. Δεν ήταν εύκολε οι συνδιαπραγματεύσει πάντοτε και με το Συμβούλιο και γι' αυτό θέλαμε να το ευχαριστήσουμε που κατάφερε ε, σε τελευταίο, ε, το δεκάτη ώρα να καταλήξει σε ένα συμβασμό. Θα ήθελα λοιπόν να ε, πω ότι θα έπρεπε και για τις δημόσιες μεταφορές, μαζικές μεταφορές να ε, συζητήσουμε το πώς θα προστατευθούν τα δικαιώματα των επιβατών. Αυτά είναι θέματα όμως τα οποία και περιφερειακά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εν γέννη υποστηρίζει λοιπόν την ε, πρόταση συμβασμού. Το βλέπουμε σε ένα πακέτο μέτρων ε, ως προς τα δικαιώματα του επιβάτη που έχουμε δει και σε άλλους τομείς των μεταφορών. Και θα θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα αργότερα να έχουμε μια κωδικοποιημένη, μια συνολική μορφή του όλου της νομοθεσίας έτσι ώστε ο επιβάτης, ο καταναλωτής ο ίδιος να έχει την επισκόπηση αυτής της νομοθεσίας και να μένει στα χέρια μόνο των ε, δικηγόρων και των δικαστών γιατί ο επιβάτης δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζει και να αναγνωρίζει τα δικαιώματά του επειδή θα είναι πολύ περίπλοκη νομοθεσία. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την πολύ καλή συνεργασία και ελπίζω ότι στην Ολομέλεια θα εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρός και τώρα θα ακούσουμε τον Brian Simpson εκ μέρου ε, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα καταρχάς ε, να εκφράσω και εγώ τις ευχαριστίες μου εκ μέρου της ομάδας μου προς τον κύριο Καντσάν για τη σκληρή δουλειά που έκανε. Πρόκειται για ένα ζήτημα περίπλοκο, δύσκολο, Είχαμε δύο κύρια ερωτήματα να αντιμετωπίσουμε, άλλωστε είναι τα πρώτα που βλέπει κανείς να εξετάζει με τέτοια συμφωνία. Πρώτο ερώτημα, είναι ιδεώδη συμφωνία. Δεύτερο ερώτημα, μας πηγαίνει προς τα μπρος, είναι βήμα πρόοδου. Για το πρώτο ερώτημα από πλευρά του Κοινοβουλίου θα απαντήσω αρνητικά. Δεν είναι ιδεώδη ε, η συμφωνία. Ο συμβασμό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αναγκάστηκε να υποχωρήσει σε κάποια σημεία, ιδιαίτερα στο πεδίο εφαρμογή, που θα θέλαμε μικρότερε αποστάσει να ισχύουν για την θέση εφαρμογή αυτή τη νομοθεσία. Για το αν αποτελεί όμω βήμα προοδού και αν μα προάγει προ τα μπρο, ναι, η απάντηση είναι ότι μπορούμε να έχουμε τώρα ε, δικαιώματα για του επιβάτε λεωφορείων και πούλμαν ισοδύναμα με αυτά που έχουν αναγνωριστεί σε άλλους ε, τρόπους μεταφορών, σε άλλα είδη μεταφορών και επίσης ταυτόχρονα βελτιώνεται και η δέσμευσή μας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε λεωφορεία και πούλμαν σε επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα ή ακόμη και επιβάτες με αναπηρίες ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα εδώ όταν ε, επί παραδείγματα γίνεται λόγος για κατάρτιση προσωπικού ε, για την ε, δυνατότητα το προσωπικό να ενημερώνεται για το πώς θα χειρίζεται και πώς θα διευκολύνει επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα ή με αναπηρίες σε αυτό το θέμα θα ήθελα να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες από κράτη-μέλη αυτή η πρόταση να καθυστερήσει για μια πενταετία ακόμη. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Και πάντως θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τελική συμφωνία ώστε τα δικαιώματα όλων των επιβατών ε, από όλους τους χώρους των από όλο το χώρο των μεταφορών να ε, θεσπιστούν και να ισχύουν κατά ομοιόμορφο τρόπο. Ίσως χρειαστεί μεταρρύθμιση αργότερα, αλλά πάντως έχουμε ε, σημειώσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου στον τομέα αυτό και ελπίζω το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει με μέγιστη πλειοψηφία το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής που επεξασφάλισε ο κ στη συνεργασία με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνερ εκ μέρου των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών. Κυρία Μάισνερ, χωρίς μικρόφωνο. Πρόεδρε, είχαμε μια μακρά διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Αυτή ήταν και η καλή είδηση. Καλή είδηση και καλή θετική πτυχή ήταν επίσης το ότι έχουμε να κάνουμε με βασικά δικαιώματα και δικαίωμα για πρόσβαση και ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και των επιβατών με περιορισμένη κινητικότητα. Επίσης έχουμε να κάνουμε με θετική είδηση όταν μιλούμε για τη δυνατότητα επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ή επίσης θετικό είναι το γεγονός ότι αν δεν είχαμε καταλήξει σε συμφωνίες στην διαλλαγή, αυτός ο τομέας των μεταφορών θα είχε μείνει έξω από τη ρύθμιση ως προς τα δικαιώματα των επιβατών. Μίλησα για τα θετικά λοιπόν στοιχεία, αλλά ασφαλώς υπάρχουν και τα αρνητικά, ότι δηλαδή στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, στον τομέα της ε, παροχής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης για τα άτομα με αναπηρίες και με περιορισμένη κινητικότητα δεν ε, καλύπτονται ικανοποιητικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εφόσον τρία κράτη μπορούν να βγουν έξω από την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Ε, επί παραδείγματι, και επίση ένα άλλο μέτρο το οποίο μα δυσαρεστεί είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με την παρουσία συνοδού για τα άτομα αυτά ή με την ε, δυνατότητα να αρνηθεί η επιχείρηση την αποζημίωση σε περίπτωση ανωτέρα βία, η οποία δεν ισχύει φερρυπίν για τι αεροπορικέ μεταφορέ γιατί στην περίπτωση του, της τέφρα είχαν υποχρεωθεί οι ε, ε, αεροπορικέ εταιρείε να αποζημιώσουν τους επιβάτες τους παρότι πρόκειται για ανώτερα βία. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν πρέπει να επανεξεταστούν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λιχτινμπέργκερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπορεί να και η σχετική σύμβαση συνθήκη. Πλην όμως τα δικαιώματα για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και περιορισμένη κινητικότητα στο θέμα αυτό δεν προστατεύονται επαρκώ. Και το λέω αυτό ξεκινώντα την παρέμβασή μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το κυριότερο έλλειμμα τη νομοθεσία αυτή. Ότι δηλαδή πάντα εισάγουμε περιορισμού στην προστασία των δικαιωμάτων με τη διατύπωση εφόσον είναι δυνατόν. Και πρέπει να πω ότι δυστυχώ εγώ γνωρίζω αρκετά καλά αυτή την κατάσταση, ώστε να είμαι σε θέση να σα διαβεβαιώσω ότι το εφόσον είναι δυνατόν ω φράση σημαίνει απλούστατα ότι δεν πρόκειται να καταστεί δυνατόν για τον επιβάτη με περιορισμένη κινητικότητα ή με αναπηρία να προβλεφθούν λύσει αποτελεσματικέ και ουσιαστικέ. Και ιδιαίτερω θα ήθελα να πω ότι αυτό περιορίζει ιδιαίτερω τον τρόπο με τον οποίο θα προσφέρεται η πληροφορία μέσα σε ένα λεωφορείο ή πούλμαν για τον επιβάτη αυτόν. Ακόμα και εδώ πέρα βλέπουμε αποδυνάμωση τη σχετική ρύθμιση Άρα δεν μπορεί να γνωρίζει ο επιβάτης με περιορισμένη κινητικότητα πού μπορεί να στραφεί για να εξασφαλίσει στήριξη και ε, βοήθεια η ενημέρωση. Επίσης ένα άλλο ζήτημα που είναι σχετικό με τις ε, τελικές αυτές, το υλικό αυτό γύρω διαπραγματεύσεων ε, των οποίων με πολύ σκληρό αγώνα ο κύριος ε, Μάντσιαν ε, προώθησε, αλλά δυστυχώς προσέκρουσε στην σκληρότητα του Συμβουλίου και δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Ήταν αυτός, όπως είπα, της ενημέρωσης και κατάρτισης των ατόμων με ε, περιορισμένη κινητικότητα, ε, το ζήτημα των 250 χιλιόμετρων που τελικά θα οδηγήσει στο να ε, κατακαιρματίζονται τα δρομολόγια, δηλαδή θα βρουν τη λύση οι επιχειρήσει αυτέ των μεταφορών, κόβοντα το δρομολόγιο στα δύο. Ένα δρομολόγιο των 500 χιλιόμετρων θα μετατραπεί σε δύο δρομολόγια των 250, προκειμένου να καταστρατηγήσουν τις διασχετικές διατάξεις και να απαλλαγούν από την υποχρέωση ενημέρωσης αποζημίωσης και Τώρα πιστεύω ότι ε, εφόσον υπάρχει η αρχή της κατάρτισης για το προσωπικό τουλάχιστον ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά κατά τα άλλα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν βλέπω να έχουμε επιτύχει κανένα μεγαλούργημα, κανένα ε, έργο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τσίλεκ μέρους των συντηρητικών μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ όλους όσους ε, συμμετείχαν στην εκπόνηση της συμβαστικής ε, λύσης ε. και συγχαίρω τον εισηγητή γιατί κατάφερε να καταλήξει στην βέλτιστη συμβαστική λύση σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Πρόκειται για τα δικαιώματα των επιβατών που κατοχυρώνται για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα επίπεδα προστασίας ανάλογα με το μέσο μεταφοράς. Οι προθεσμίες για την αποζημίωση, ό,τι προβλέπεται για τις ματαιώσεις, για τις καθυστερήσεις. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές διατάξεις, όπου και μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση τους καταναλωτές. Πάντως, ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση και μεριμνούμε ώστε να εφαρμοστεί μια επαρκής προστασία για τους καταναλωτές και το ότι καταλήξαμε στη συμβαστική λύση τελευταία στιγμή είναι αυτή απόδειξη της δυσκολίας ε, του ζητήματος. Ε, κατόπιν για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ε, είναι ικανοποιητικές οι ρυθμίσεις ε, και ε, προφανώς θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για αποστάσεις σε μικρότερες των 250 χιλιόμετρων. Συμφωνώ επίσης με τα σχόλια που ακούσαμε ως προς την ενημέρωση των καταναλωτών ε, και δεν με ικανοποιεί η παρέκκληση που έχει χορηγηθεί στις, στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε. της κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συναδελφοί, τα δικαιώματα των επιβατών ε, σε όλα τα μέσα μεταφοράς είναι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Ομολογώ ότι διακρίνω κάποια προβλήματα που ενδέχεται ε, να προκύψουν. Παραδείγματος χάρη... μπορεί με τα θεσπιστέντα μέτρα να οδηγηθούμε σε αύξηση κάποιων μέσων μεταφοράς ε, και του κόστους ε, για κάποια ε, είδη μεταφοράς. Τώρα, σε σχέση με τις καθυστερήσεις και τις ματαιώσεις των δρομολογίων, Συμφωνώ με τα μέτρα που προτείνετε και θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο, την κυρία Κράτσα, τον κύριο Σίμψον, τον κύριο Κάτσεν, τον εισηγητή μας, ε, ε, γιατί είναι λογική και ρεαλιστική η λύση στην οποία κατάληξαν. Ε, λοιπόν, ας πάρω τα θετικά σημεία. Είπαμε, απόσταση άνω των 250 χιλιόμετρων και αυτό θα καλύπτει και τους επιβάτες που διανύουν μόνο ένα τμήμα αυτής της απόστασης. δεύτερον, αναβαθμίζεται η κατάσταση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα Τρίτον, ε, αποζημίωση και αρρωγή σε περίπτωση ατυχημάτων. Ε, επ' αυτού θα ήθελα να πω ότι ε, όταν υπάρχει κάποια ζημία, προβλέπετε ότι θα υπάρξει αποζημίωση στο ακέραιο. Παραδείγματο χάρη για τι αναπηρικέ ε, καρέκλε. Νομίζω ότι σε κάποιες ε, περιπτώσεις ε, θα πρέπει να επιδιώξουμε ανώτερα ωραία και κυρίως ε, να επιδιώξουμε σωστή ενημέρωση των καταναλωτών. Πέμπτον, ε, καλωσορίζω την μεταβατική περίοδο. Έχει μειωθεί στα τέσσερα χρόνια. Βεβαίως ε, δυσαρεστήθηκα διότι βλέπω πιθανότητα ε, ανανέωσης της μεταβατικής περίοδου. Επίση, χαίρομαι που καλύπτονται οι επιβάτε που διανύουν ένα μόνο κομμάτι τη απόσταση Τώρα για τα οικονομικά όρια, τα όρια αποζημιώσεων, δεν λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός ε, ε, ούτε και η ισοτιμία ε, του ευρώ. Πάντως, εν γέννη είναι πολύ καλή συμβαστική λύση και όλες οι προσπάθειές που θα πρέπει να κατευθύνονται προς την αυξημένη προστασία των επιβατών. Η ομάδα μας υποστηρίζει λοιπόν την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ιμπράσας από την Ένωση για την Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι. Διότι μετά από μακρά συζήτηση και διαπραγμάτευση, το κείμενο που έχουμε ενώπιόν μας μπορεί να θεωρηθεί ε, ένας πολύ καλός συμβιβασμός, διότι επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των ε, επιβατών χωρίς να επιβαρύνει τους ε, φορείς αυτούς. Εάν λάβουμε υπόψη την ευρύτερη πρόταση περιλαμβάνει πολύ μεγαλύτερα και ευρύτερα δικαιώματα σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφοράς και δίνει ίσους, εξασφαλίζει ίσους όρους πρόσβασης στα κράτη-μέλη. Αυτός ο κανονισμός ορίζει ότι οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν σε περίπτωση ε, τραυματισμού, ε, απώλειας, απώλειας ή ζημίας των αποσκευών εξαιτίας ατυχήματος και σε περίπτωση θανάτου. Επίσης θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη αρρωγή σε περίπτωση ατυχήματος, δηλαδή παροχή ε, τροφής και ρουχισμού. Αν υπάρξει καθυστέρηση άνω των 120 λεπτών, μπορεί να ε, λάβει αποζημίωση που θα ισούται με 50% της, ισίας του, της αξίας του εισιτηρίου ο επιβάτης. Και αυτό αφορά και τα δικαιώματα ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Ο επόμενος ομιλικής, ο κύριος Όπερμαϊερ. Υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των επιβατών... Νομίζω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον δύο διανυκτερεύσεις ε, για μια καθυστέρηση ε, ή ματέωση ταξιδιού για τον επιβάτη. Υπάρχουν όμως διάφοροι παράγοντες που δεν μπορεί να επηρεάσει η ίδια η εταιρεία. Όταν, παραδείγματι, παράδειγμα δυσμενείς καιρικές συνθήκες ε, ή όταν δεν υπάρχει η πετιότητα της επιχείρησης για κάποια καθυστέρηση ή ματέωση. Το ίδιο νομίζω θα πρέπει να δούμε και στις δρομικές μεταφορές, όπως επίσης καθυστερήσεις σε ε, λεωφορεία που δεν έχουν προξενήσει τα ίδια. Φερρυπίν στις αστυνομικές ε, μεταφορές όταν έρχεται ένα τρένο από τη Γερμανία προς την Αυστρία με μεγάλη καθυστέρηση λόγω όμως των γερμανικών σιδηροδρόμων δεν μπορεί να θεωρηθεί ω υπέτεια η αυστριακή επιχείρηση σιδηροδρόμων. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα λεωφορεία. Ευχαριστώ πολύ λέει η πρόεδρο. Έχουμε τώρα τον κύριο Κόχ. Είναι ομιλητές εξ παρακαλώ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ που δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, απόφαση τη Επιτροπή Συνδιαλλαγή. Θα μπορέσουμε και στον τομέα των λεωφορείων και πούλμα να εξασφαλίσουμε υψηλέ προδιαγραφέ προστασία για του επιβάτε, αντίστοιχο με αυτό που έχουμε και σε άλλε μεταφορέ. Για άλλου του επιβάτε, λοιπόν, και εκείνου που έχουν περιορισμένη κινητικότητα. Και δεύτερον, μπορούμε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών. Και τρίτον, μπορούμε να έχουμε ε, μια ιδιαίτερη μεταχείριση σε περιπτώσεις ε, που έχουν να κάνουν, ε, μάλλον στον τομέα αυτών που έχει πιο πολύ γνωρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορέσαμε ε, προτάσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν ως εφαρμόσιμες να τις ε, βγάλουμε από την πρόταση και έτσι να έχουμε μια καλή συμβαστική λύση. Πρέπει οι άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα αναπηρίας ή κινητικότητας να έχουν δικαίωμα και σε παροχή βοήθειας για λόγους και κοινωνικής ενσωμάτωσης δωρεάν. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σερακιάνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Καντσάν για τη δέσμευσή του έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτός ο συμβιβασμός διότι έτσι οι επιβάτες των οδικών μεταφορών μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με επιβάτες σιδηροδρόμων ή πλοίων. Μιλάμε για απόσταση που ισούται ή υπερβαίνει τα 250 χιλιόμετρα και βεβαίως μιλάμε και για επιβάτες μικρότερων ε, αποστάσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. Θα μπορέσουν να ε, αποζημιώνονται ε, εάν υποστούν ζημία τα αναπηρικά αμαξίδια τους. Επίσης μιλάμε και για αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου συμπεριλαμβανομένων λογικών εξόδων κηδείας ή σε περίπτωση προσωπικού τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας των αποσκευών εξαιτίας ατυχήματος. Επίσης, εάν ε, έχουμε ε, ματαιώσεις ή καθυστερήσεις, η αποζημίωση του ε, επιβάτη θα ισούται με 50% της αξίας του εισιτηρίου. Παράλληλα με την επιστροφή της τιμής εισιτηρίου. Τέλος, χαίρομαι διότι για τα άτομα με ανεπηρία και με μειωμένη κινητικότητα θα εγγυηθούμε την καλύτερη δυνατή αρρωγή και να μπορέσουν να έχουν ένα συνοδό ο οποίος να μην ε, επομίζεται έξοδα μεταφοράς. Η κυρία Μπιλμπάου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καντσάν, ο οποίος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει σε αυτό το, το επίτευγμα. Μιλήσαμε για τα δικαιώματα επιβατών ως προς την αποζημίωση σε περίπτωση ματέωση καθυστέρησης, σε περίπτωση ατυχήματος και ε, τα δικαιώματα ατόπων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα ανεξάρτητα από την ε, απόσταση. Νομίζω όμως ότι τη στιγμή που μιλάμε για 250 χιλιόμετρα αποκλείονται τρεις χώρες. Κατανοούμε ότι επιτεύχθη προόδος σε σχέση με το αρχικό ε, προτινόμενο, αλλά θα απόσχουμε. Ο κύριος Τσαρνέτσκι για 1,5 λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστέλει ένα πολύ βασικό θετικό μήνυμα στους επιβάτες, στους φορολογούμενους και στο εκλογικό μας σώμα. Όλους δηλαδή που χρησιμοποιούν λεωφορεία και πούλμαν και ε, τα άτομα με αναπηρίες ή με μειωμένη κινητικότητα χρειαζόμαστε τέτοιες απτές αποφάσεις διότι οι φορολογούμενοι καταβάλουν το αντίτιμο και αυτοί μας πληρώνουν, καταβάλουν δηλαδή και τους μισθούς μας σε τελευταία ανάλυση. Βεβαίως δεν είναι ιδεατή αυτή η νομοθεσία αλλά νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ανθρώπινη και πιο ανοιχτή για τις ανάγκες όχι των πολιτικών, αλλά των καταναλωτών των κοινών Ευρωπαίων. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Καντσάν για την εξαιρετική ε, αυτή έκθεση. Ρόσπαχ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι βοηθάμε τους επιβάτες και στην περίπτωση καθυστερήσεων ή ματαιώσεων. Αυτό είναι πολύ καλό. Θα ήθελα όμως να επικρίνω το εξής. Αυτό που μετράει ιδιαίτερα είναι τα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. Όμως τα λεωφορεία δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή για να μεταφέρουν άτομα με μειωμένη κινητικότητα ε, επίσης ως προς το αντίτιμο των εισιτηρίων ε, έχει πέσει αρκετά για να υπάρχει ανταγωνιστικότητα με τις εναέριες μεταφορές. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο οι αποζημιώσεις θα μπορέσουν να καταβληθούν από τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να κλείσουν σε περίπτωση καταβολής ε, μεγάλων αποζημιώσεων. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τις ΜΜΕ περισσότερο. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπαχ ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους ε, τους συναδέλφους, ιδιαίτερα τον κύριο Κάντσαν για τις προσπάθειές τους και τους σκληρούς αγώνες για την εξέβρεση συμβασμού σε αυτό το δύσκολο θέμα. Υπήρξαν ήδη επιτυχίε που ακούστηκαν, αλλά και αποτυχίε, όπω η παραδειγματή το πεδίο εφαρμογή και διάφορα άλλα σημεία, ε, τα οποία δυστυχώ δεν ε, πετεύχθησαν. Έχουμε, πιστεύω, καλύψει με το νέο αυτό μέτρο όλους τους τομείς των μεταφορών και τα δικαιώματα των επιβατών και τώρα το επόμενο βήμα θα είναι να έχουμε μια κωδικοποίηση, μια ενοποιημένη νομοθεσία ορατή για τον καταναλωτή και επιβάτη. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τον ε, πολίτη και πάνω απ' όλα η συνοχή του δικαίου θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή διαφορετικά κριτήρια Όλο διόλου διαφορετικά κριτήρια για τον επιβάτη αεροπορική εταιρεία σε σχέση με αυτά τα οποία ε, προβλέπει νομοθεσία για τον επιβάτη ε, νέας επιχειρήσης ε, οδικών μεταφορών και σεών μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σελκαντράου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα Φυσικά να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή, το, του σκιώδη εισηγητές, τον κύριο Σίμψον, την κυρία Κράτσα, όλου όσου κατέβαλαν προσπάθειε για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Προφανώς ευχαριστώ και την Βελγική Προεδρία. Θα ήθελα να είμαι λίγο επικριτικός ενώπιον του Συμβουλίου. Λυπούμε που το πεδίο εφαρμογή καλύπτει αποστάσεις ίσες ή άνω των 250 χιλιόμετρων, ενώ με τα ευρωπαϊκά δεδομένα θα ήταν λογικό Όλε οι διασυνοριακέ μεταφορέ να εμπίπτουν στο στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Τα 250 χιλιόμετρα ε, δεν, έτυχε, ε, δεν έτυχαν τι υποστηρίξει όλων των κρατών μελών καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία ε, και σε αυτό το αμφιλεγόμενο ζήτημα κατέστη πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μια πλειοψηφία κρατών μελών που έχουν ω βασική μεριμνά του την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών. Ο κανονισμός αυτός ε, μας επιτρέπει, ε, μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε την εξέταση του ζητήματος, καλύπτοντας όλα τα μέσα μεταφοράς ε, και ο Επίτροπος ήδη προανήγγειλε πως θα ξεκινήσει το πείραμα οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να εφαρμοστούν και κατόπιν να αποτιμήσουμε την ε, θέση σε εφαρμογή τους. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί βασικά δικαιώματα πλέον σε επιβάτε ε, πούλμαν και λεωφορείων. Έχουμε προβλέψει αποζημιώσει ε, σε περίπτωση σημαντικών καθυστερήσεων ή ματαιώσεων δρομολογίων, καθώς και αρρωγή για τους επιβάτες που το χρειάζονται η συμβαστική λίστα τεθεί σε ισχύ σε δύο χρόνια, προβλέπεται μεταβατική περίοδο πάντω είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση και είναι μια ε, καλή ισορροπία ανάμεσα στι υψηλέ φιλοδοξίε του Κοινοβουλίου και τη μετριοπαθή στάση του Συμβουλίου Αφετέρου. κυρία Σάβησαρ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Λένε οι Εσθονοί ότι όταν αφιερώνουμε πολύ χρόνο σε κάτι το αποτέλεσμα είναι καλό έχουμε μια σχετική λαϊκή ρίζη. Δυστυχώ δεν μπορώ να ισχυριστώ το ίδιο ως προς τον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών. Η διαδικασία συνδιαλλαγής ε, ήταν ατέρμονη και κατά τη διάρκεια αυτή τη διαδικασία απομακρυνθήκαμε από τις αρχές ε, των οποίων υπεραμεινόταν ε, το Κοινοβούλιο. Έχουμε κάποια βασικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον κανονισμό, πλην όμω η απόσταση ίση ανώτερη των 250 χιλιόμετρων ε, αποκλεί ε, από το πεδίο εφαρμογή τρει χώρε και πέρα από αυτέ τι ε, τρεις χώρες υπάρχει και μία χώρα για την οποία καλύπτεται ένα τμήμα μόνο των δρομολογίων. Ε, κατόπιν ε, οι διασυνοριακές ε, τακτικές γραμμές ανεξαρτήτως απόσταση θα έπρεπε να καλυφθούν. Δεν μπορούμε να δεχθούμε την εξαίρεση αυτή. Η εστονική κυβέρνηση δυστυχώς υποστήριξε τους όρους και αξίωνε μία μεγαλύτερη απόσταση μάλιστα. Ε, υποστηρίζουμε τελικά τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών ή ε, υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των παρόχων, των μεταφορικών εταιριών. Εγώ είμαι με το μέρος των επιβατών και δεν κατανοώ πραγματικά γιατί αποκλείουμε από αυτόν τον κανονισμό ένα κομμάτι της Ευρώπης. Πρόεδρος, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να σα το υπενθυμίσω. Ο κύριο Μπράντμπορν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω πλήρως ε, τα δικαιώματα των ε, επιβατών. Ε, είναι λογικό να περιμένουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και υπηρεσιών οι κατάλληλες. Αλλά πρέπει να τηρούμε και τις αναλογίες. Δηλαδή, ποιες συνέπειες θα έχουν αυτά τα μέτρα. Να συγκρίνουμε τα πραγματικά ωφέλη για τους καταναλωτέ, με το πραγματικό κόστος που συνεπάγεται αυτό για τον κλάδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μια ομοιόμορφη λύση. Όμως τα δικαιώματα των επιβατών ποικίλουν ανάλογα με το μέσο μεταφοράς. Άλλο αεροπλάνο, άλλο ε, πούλμαν, άλλο λεωφορείο. Εδώ μιλάμε για μικρομεσαίε επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα και πιστεύω ότι όλοι γνωρίζονται πόσο σημαντικό είναι να είναι αξιόπιστε οι υπηρεσίε και πόσο σημαντικό είναι αυτό για τι τοπικέ ε, οικονομίε όταν μιλάμε για τους, ε, τα πούλμαν και τα λεωφορεία. Η απόσταση τώρα των 250 χιλιόμετρων μα είναι άδικο για τι εγχώριε μικρέ επιχειρήσει που προτείνουν, προσφέρουν συγγνώμη, τοπικά δρομολόγια να μην καλύπτονται από το κανονικό. Υποστηρίζω παρόλα αυτά τον γενικότερη συμβαστική λύση λόγω των θετικών σημείων της. Ο κύριο Χίγκιν, ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ και τρία χρόνια σχεδόν ε, οφορούμε αυτή την πρόταση και ε, για πρώτη φορά μάλλον τάσσομαι με το ε, Συμβούλιο παρά με το Κοινοβούλιο. Φυσικά θέλουμε να προστατεύσουμε τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, αλλά όπως είπε ο Φίλιπ Μπράντμουν, αν εγκριθούν αυτές οι προτάσεις, οι μικρές εγχώριες επιχειρήσεις δεν θα επιβιώσουν, θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα. Γι' αυτό και ήταν τόσο σημαντική η συνδιαλλαγή και η συμβαστική λύση, νομίζω, οδηγεί σε μια ισορροπημένη λύση ανάμεσα στα συμφέροντα των παρόχων υπηρεσιών και τα αφενός και των δικαιωμάτων καταναλωτών αφετέρου. Ε, σχετικά με τα δικαιώματα τώρα, είτε μιλάμε για αεροπερορικές ε, και συνδρομικέ ε, και οδικές μεταφορές, δεν μπορούν να είναι τα ίδια, εξαρτάται από το μέσο μεταφοράς, δεν μπορούμε να έχουμε ένα νέο πακέτο, δεν είναι εφικτό, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Μπρέιαν Σίμψον, τον πρόεδρο τη Επιτροπή Μεταφορών, εργάστηκε εξαιρετικά. Ε, συγχαίρω τον εισηγητή, κύριο Κιάνκεν, ε, τον δικό μα συντονιστή και ευελπιστώ ότι ε, τελικά θα καταλήξουμε σε ένα ε, υποφέλε για όλου συμβαστικό πακέτο. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Φλασάκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, στο παρελθόν ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν διατάξει σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις εναέρειες και δρομικέ μεταφορές. Είναι ως εκ τούτου λογικό να εγκρίνουμε έναν παρεμφερή κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών πουλμαν και λεωφορείων. Οι επιβάτες ε, στην Ευρώπη προτιμούν τις κάποιες ε, μετακινήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών. Ε, χρειάζεται να θέσουμε όρια, κυρίω σε σχέση με τις διασυνοριακές ε, μεταφορέ και ω προ τι ευάλωτε πληθυσμιακέ ομάδε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους. Ε, δεν είναι σωστό να επιβάλλουμε αυτά τα δικαιώματα σε μικρές ε, τοπικές επιχειρήσεις ή να ισχύουν για πολύ μικρές αποστάσεις. Η υπερβολική κανονιστική ρύθμιση συνιστά άχθος για, τους, ε, για τις μεταφορικές εταιρείες ε, όπου θα οδηγήσει σε αύξηση των άβλων των εισιτηρίων, των δρομολογίων. Οι τοπικέ ε, μεταφορικέ εταιρείε λοιπόν είναι καλό να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογή των κανονισμών, ώστε να μην είναι υπερβολικέ οι νομοθετικέ διατάξει. Ήταλα. Για ένα λεπτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό τον συμβασμό και ιδιαίτερα τον εισηγητή και τον κύριο Σίμψον. Βεβαίως είναι συμβιβασμός αλλά είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός ενώπιον του πολίτη. Ιδιαίτερα να λάβουν υπόψη περιπτώσεις ατυχημάτων ή καθυστηρήσεων ή ε, αποσκευών που χάνονται. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει προστασία των ε, επιβατών. Βεβαίως τα 250 χιλιόμετρα δεν είναι η καλύτερη δυνατή διευθέτηση. Νομίζω ότι είναι ο πιο αδύναμος κρίκος αυτής της νομοθεσίας και θα πρέπει να επανέλθουμε αργότερα. η τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα έχουν ε, περισσότερα δικαιώματα. Τέτοια δικαιώματα θα πρέπει να προωθούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτή η, ε, η διάταξη είναι πολύ καλή, αλλά μόνο ως προς ορισμένα μέρη, δηλαδή ως προς ορισμένους θύλακες. Και αυτό αφορά τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη ε, κινητικότητα. Μιλάμε όμως για 250 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί να ισχύει ένας νόμος για όλους. Στα 27 κράτη-μέλη θα έπρεπε να υπήρχε μια ευελιξία μέσα στις χώρες έτσι ώστε όλες να μπορούσαν να συμπεριληφθούν. Εγώ πρέπει να διανύσω 300 χιλιόμετρα και στη δική μου εκλογική περιπτώση μέχρι να φτάσω το Δουβλίνο θα πρέπει να διανύσω 300 χιλιόμετρα και τώρα θα υποστούν μεγάλη πίεση αυτοί οι μεταφορείς και μέσα στα πλαίσια της καταβολής ασφαλίστρων, διότι θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας και επίσης πολλές διευκολύνσεις των επιβατών που θα χαθούν. Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία Catch the Eye Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων. Ο κύριος Κόζα έχει το λόγο. Θα πρέπει να μιλήσουμε μόνο πέντε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες με ε, αναπηρίες μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνεται και να διεκδικήσουν την εφαρμογή την, ε, το σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες θα πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστά χωρίς κανένα πρόσχημα για περιορισμό τους. Δυστυχώς όμως το Συμβούλιο δεν ήταν τόσο ακέραιο σε αυτή την θέση και δυστυχώς δεν αναγνώρισε πλήρως αυτά τα δικαιώματα το, Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο ε, των Υπουργών. Ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε για τον κάθε πολίτη της Ευρώπης την δυνατότητα αυτή. Γιατί κάθε μέρα υπάρχουν περισσότεροι πολίτες με αναπηρίες, με περιορισμένη κινητικότητα και ο κάθε πολίτης ανα πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί σε αυτή την θέση. Πρέπει λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε μετά τη συμβαστική ε, ρύθμιση να στην υλοποίηση και τον ουσιαστικό σεβασμό των δικαιωμάτων των επιβατών με αναπηρία. Ευχαριστώ κυρία Συναλόβα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε αυτό το σημαντικό συμβασμό, ο οποίος ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών σε λεωφορεία και πούλμαν και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονό ότι προσφέρεται δυνατότητα για αποζημίωση σε καθυστερήσεων, ματαιώσεων ή ατυχημάτων με ιδιαίτερη με έρημνα για τα άτομα με αναπηρίες ή με κινητικά προβλήματα. Ιδιαίτερη δε σημασία δίνω στην ε, θεματολογία της σχετική με την ενημέρωση των επιβατών ε, και την παροχή βοήθειας ε, που συζητήθηκε στην συνδιαλλαγή. Δεν ήταν εύκολο να εξασφαλιστεί συμβασμό, το γνωρίζω και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι ενεπλάκησαν στην διαδικασία της συνδιαλλαγής. Με τον κανονισμό αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε η ικανοποιητική και ισότιμη κάλυψη των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφορών. Μπορεί να μην είναι τέλεια η κατάσταση, αλλά προχωρεί προς το καλό σκοπό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρίση έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα απόσχουμε τη, στην ψηφοφορία και όλοι οι φιλελεύθεροι για τον κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών πούλμαν και λεωφορείων. Είναι το τελευταίο κομμάτι τη ολισίδα μετά τη, τα αεροπλάνα, τα πλοία για τα τρένα. Είναι πολύ λιγότερο πρόταση. Το ακούσαμε αυτό. Από τους σοσιαλιστές ακούσαμε τον κύριο Σίμψον και τον κύριο Χαντράουι. Το ανέφεραν. Η απόσταση των 250 χιλιόμετρων δεν συνιστά επαρκή προστασία. Ε, δηλαδή, ε, ε, μπορείτε να καλυφθεί Ηταν αν κάνετε ε, το Άμστερνταμ Βρυξέλλες ε, με αεροπλάνο, αλλά όχι αν το κάνετε με ε, πούλμαν. Οπότε είναι σε πλεονεκτική θέση κάποια μέσα μεταφορά. Σχετικά τώρα με τις αποκλήσεις, το 2012 θα αρχίσουν να ισχύουν τα δικαιώματα αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης, αιματέωσης κτλ. Μα χρειαζόμαστε αυτή την βοήθεια, κυρίως για τα μειονεκτικά άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Σίγουρα δεν θα εφαρμοστούν και τα γρήγορα τα μέτρα και σίγουρα όχι για όλους. Ευχαριστούμε κύριος Κρέιμερ. Πολύ καλό είναι το ότι συζητούμε τώρα ισότιμη μεταχείριση και δικαιώματα για τους επιβάτες σε όλα τα είδη των μεταφορών, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας κάνει το γεγονό ότι ο σιδηρόδρομος που είναι και το πιο οικολογικό μέσο μεταφοράς έχει μειονεκτική ε, έχει διακριτική μεταχείριση, επιβαρύνεται δηλαδή με πολύ ψηλότερη αποζημίωση για μικρότερη απόσταση σε σχέση με το λεωφορείο. Μειονέκτημα λοιπόν για τον σιδηρόδρομο ε, πλεονέκτημα για το λεωφορείο και το πούλμαν. Ε, στη μία ώρα καθυστέρηση ο σιδηρόδρομος, το, η σιδηροδρομική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση, ενώ χρειάζεται να έχει καθυστέρηση δύο ώρων στα, στις ε, οδικές μεταφορές ε, η επιχείρηση λεωφορείων για να αποζημιώσει τον επιβάτη. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει τόσο διακριτική μεταχείριση. Πολλά έχουμε ακόμα να κάνουμε λοιπόν και δεν είναι καλός αυτός ο συμβασμός των 250 χιλιόμετρων. Ενώ για το, οι σιδηροδρομικές μεταφορές κάθε τρένο ε, έξω από τις πόλεις, περαστικό δηλαδή, θα καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση ε, καθυστερήσεων. Ευχαριστώ κύριος Πάσκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ύστερα από περίπλοκες ε, διαπραγματεύσεις και συνδιαλλαγή καταλήγουμε, Πρόεδρε, σε μια συμφωνία για τα δικαιώματα των επιβατών σε λεωφορεία και πούλμαν. Και και ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ε, δρομολόγια τουλάχιστον 250 χιλιόμετρων, πιστεύουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με σημαντικό βήμα για την προστασία των καταναλωτών, επιβατών, σε περιπτώσεις δηλαδή καθυστερήσεων, ε, επιβάλλεται η επιστροφή ακέραιου του εισιτηρίου ή και αποζημίωση 50%. Το πρόβλημα είναι εκεί όπου υπάρχουν παρεκκλήσεις από το προσορισμένο χρονοδιάγραμμα που σημαίνουν ότι ορισμένα μπορούν να καθυστερήσουν για 4 συν 4-8 χρόνια το συνολικό διάστημα θέση εφαρμογή των διατάξεων. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Επίτροπος, Επίτροπος παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι βουλευτές για τα πολύ θετικά καταπλειονότητα σχόλια. Τώρα προχωρούμε στη μεγάλη πρόκληση της υλοποίησης της ουσιαστική εφαρμογής αυτής της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών στις χερσαίες μεταφορές και βεβαίως έχουμε ένα διάστημα μπροστά μας στο οποίο θα χρειαστεί να διευκρινίσουμε κάποια στοιχεία συγκεκριμένα της νομοθεσίας αλλά νομίζω ότι ο συμβασμός που θα υιοθετηθεί πιστεύουμε αποτελεί μεγάλο κείμενο και εξυπηρετεί αρχές σημαντικές. Αρχές σημαντικές που εισαγάγαμε με την νομοθεσία αυτή στον τομέα των μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν, αρχές που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των επιβατών, ναι, έστω οι συμβασμοί είναι λιγότερο φιλόδοξοι από ό,τι θέλαμε. Ναι, έστω οι συμβασμοί πρέπει να προχωρήσουν και σε υλοποίηση ουσιαστική. Αλλά παρόλα αυτά ελπίζω ότι θα υπερψηφίσετε τον κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εξ ονόματος του Συμβουλίου, κυρία Γκόρη. Κύριε Ισήγητα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις για αυτή τη συζήτηση που μόλις διεξήχθη φάνηκαν οι δυσκολίες και τα προσκόμματα και φαίνεται που θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη, όπως φάνηκε και στην διαδικασία της συνδιαλλαγής. Πιστεύω ότι αυτό το πακέτο δεν είναι το καλύτερο δυνατό σε σχέση με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν. Όμως το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Η κατάσταση θα βελτιωθεί όταν τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο κανονισμός. Και οι απαντήσεις θα είναι πιο σαφείς. Πιστεύω λοιπόν ότι οι επιβάτες θα έχουν καλύτερη κάλυψη στο μέλλον, αν και ένα συμβιβασμό είναι πάντα συμβιβασμός. Υπάρχουν ε, δύσβατα ζητήματα όπου θα πρέπει να βρεθεί ένας κοινό τόπος. Εδώ καθίσταται πρόδειλο από όλες τις παρεμβάσεις ότι θα πρέπει να ορίσουμε, να θέσουμε ένα ορόσημο για την προστασία των ΜΜΕ, διότι θα πρέπει μας, να μας απασχολήσει η βιωσιμότητά τους. Όμως δεν μπορούμε να ξεχνάμε τα δικαιώματα των επιβατών που είναι πρώτη τη σημασίας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή προστασία για τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα. Και πιστεύω ότι αυτό το τμήμα του κανονισμού είναι πολύ καλά καταρτισμένο. Και πιστεύω ότι αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Η Ουγγρική Προεδρία πιστεύει σε μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση που να δίνει περισσότερα, να εκχωρεί περισσότερα δικαιώματα στους επιβάτες και στους πολίτες που είναι το επίκεντρο όλων των μελημάτων μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι επιβάτες και οι πολίτες έχουν μεγαλύτερα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ όλους για την εργασία αυτή και νομίζω ότι αυτό το έγγραφο μπορεί να εγκριθεί χωρίς πρόβλημα. Και τώρα δίνουμε το λόγο στον κύριο Καντσάν, στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν και εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται για τον καλύτερο δυνατό κανονισμό, αλλά ήταν και ο μοναδικός δυνατός, λαμβάνοντας υπόψη την άτεγκτη θέση του Συμβουλίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι πιστεύω ότι είτε για τις μεταφορές είτε για τον τουρισμό θα πρέπει να βρούμε μία ισορροπία και γι' αυτό το μέσο μεταφοράς μια ισορροπία η οποία θα εγγυάται την βιωσιμότητα των ΜΜΕ που θα πρέπει να τις διασώσουμε γιατί έγινε λόγος επιμακρών για αυτό το θέμα. Επίσης, ως προς τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους ή τα άτομα με πρόσκαιρη μειωμένη κινητικότητα, θα πρέπει να μην υπάρχουν διαφορές. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Και εδώ προσπαθήσαμε να επιφέρουμε μία ισορροπία που νομίζω καταφέραμε με τη συνεισφορά όλων. Νομίζω ότι ο κύριος Κάλλας μιλά για έναν ενιαίο κανονισμό για όλα τα μέσα μεταφοράς και τη δημιουργία ε, μιας ενιαίας αγοράς των μεταφορών. Κάτι το οποίο δεν είχαμε επιτύχει μέχρι τούδε, ιδιαίτερα ως προς την εποπτεία των δικαιωμάτων των επιβατών. Θα πρέπει να υπάρχει και ένας οργανισμός αναφοράς και ένα ενιαίο εισιτήριο για, όλες τις, ε, για, όλους, για όλα τα μέσα μεταφοράς. Ευχαριστώ τους Κιώδης και όλους όσους συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην τελική διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ την Επιτροπή Τραν και το προσωπικό και τη γραμματεία, καθώς και την Ουγγρική ε, Προεδρία. Ευχαριστώ την ε, Υπουργό Γιώρη και τον Επίτροπο Κάλλας, ο οποίος συνεισέφερε καθώς και το προσωπικό της Επιτροπής Συνδιαλλαγής που έδειξε μεγάλο και υψηλό επαγγελματισμό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις για τους πολίτες μας. Ήταν μια πολύ καλή ε, διαδικασία συνεργασίας. Η συζήτηση έχει κλείσει και η ψηφοφορία θα λάβει ε, χώρα σήμερα στις 12.